των πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της σημερινής μας συνεδρίασης. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε την ε, Παγκόσμια ημέρα γυναικών. Η ισότητα γυναικών και ανδρών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς αυτή η ισότητα δυστυχώς μόνο στα χαρτιά υφίσταται. Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίδια δουλειά έχουν περίπου 16% μικρότερο μισθό από ότι οι άνδρες. Πλήττονται ιδιαίτερα οι γυναίκες από την κρίση, χάνουν την απασχόλησή τους και πρέπει επισφαλείς θέσεις εργασίας να, να δέχονται. Υπάρχει βία γυναικών σε απαράδεκτο μέτρο με σοβαρότατες επιπτώσεις για τις γυναίκες αυτές και όλους τους εμπλεκόμενους, τις οικογένειες και συνολικά την κοινωνία μας. Πέραν αυτών, οι γυναίκε υποεκπροσωπούνται και σε ηγετικέ θέσει και στην πολιτική και στην οικονομία. Όλα αυτά τα προαναφερθέντα στοιχεία δείχνουν ότι ο αγώνα για την ισότητα των δύο φύλων δεν πρέπει να χαλαρώσει. Επιτρέψτε μου όμω, σε σχέση με την Διεθνή ημέρα γυναικών να στρέψω την προσοχή σα σε ένα από τα πιο δραματικά προβλήματα που υφίστανται και που εγώ και πιστεύω ότι και πολλοί από εσά γνωρίζετε εξίσου πάνω από 100 εκατομμύρια γυναίκες, ιδιαίτερα κορίτσια, κοπέλες, πλήττονται από τον γενετικό ακροτηριασμό αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να δεχθεί ή να δικαιολογήσει με κανένα τρόπο. Αποτελούν πραγματικά μια επίθεση και παραβίαση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των γυναικών και της ελευθερίας των γυναικών. Είναι μια παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου που κανείς από εμά δεν μπορεί να δεχθεί και δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Τέτοιες πρακτικές πρέπει με μηδενική ανοχή να αντιμετωπίζονται από πλευρά μας. Πρέπει κατεπηγόντως να δημιουργηθούν τα σωστά μέσα και εργαλεία για να προστατεύονται τα κορίτσια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ιδιαίτερα και εκτός και στην πρακτική εφαρμογή καθημερινά πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη μάχη για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι εδώ, το ότι και εδώ πάλι σήμερα, για άλλη μια φορά, έχουμε ένα τρομερό συμβάν το οποίο έπρεπε να λάβουμε υπόψη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 7 όμοιροι στην Ιγυρία από τον Λίβανο, την Ελλάδα, την Ιταλία ε, από μια τρομοκρατική οργάνωση με, το, με το, την ονομασία Ανσάρου εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν στην Ιγυρία. Εξ ονόματός σας νομίζω μπορώ να πω ότι ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει κάθετα αυτές τις πράξεις βίας και τα συλληπιτήριά μας εκφράζονται προς τους οικείους και τις οικογένειες των θυμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κυρίες και κύριοι,